την έκθεση η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα και λυπούμε που ο κύριος Ντάλι είναι απόν για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ετσεβερία για την έκθεσή του και αύριο θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Ε, το επόμενο σημείο είναι η έκθεση της κυρίας Γκάλλο για την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά. Θα δώσω τον λόγο ε, στην εισηγήτρια. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποφεληθεί της ευκαιρίας της ψηφοφορίας αυτής της εισήγησης πρωτοβουλίας που δεν είναι η δική μου εισήγηση αλλά το αποτέλεσμα πολλών συμβιβασμών για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ και δέκα χρόνια περίπου σε όλα τα κείμενά μας επαναλαμβάνουμε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να είναι η οικονομία της γνώσης, θα πρέπει να είμαστε στο ύψος αυτής της πρόκλησης που έχει γίνει πλανητική ε, πρόκληση με την ψηφιακή εποχή. Οι επιχειρήσει οι καινοτόμες αντιπροσωπεύουν 7% του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και 14 εκατομμύρια θέσει εργασία. Είναι και πρέπει να παραμείνουν το βασικό ατού πλεονέκτημα τη ευρωπαϊκής Οικονομία απέναντι ε, σε, μια, ε, σε έναν θηριώδη ανταγωνισμό πρέπει να τις προστατεύσουμε τις θέσεις αυτές, ιδαλλιώς θα εξαφανιστούν. Ποιο είναι το εργαλείο προστασίας, ποιο είναι το μέσο το οποίο θα παρακινεί τους δημιουργούς να καινοτομούν, που θα εξασφαλίσει την ποικιλομορφία, την πολιτιστική, την ευρωπαϊκή και την διεθνή της ακτινοβολία. Ποιο μέσο επιτρέπει να μπορούμε να αμείψουμε τους δημιουργούς, τους διανοούμενους, τους καλλιτέχνες. Ποιο είναι το εργαλείο που επιτρέπει την λειτουργία και ανάπτυξη των δημιουργικών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Ποιο είναι το εργαλείο που ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες και τους νέους δημιουργούς να επιχειρούν και να μεταμορφώσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μέχρι το 2020. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι προφανής. Ε, είναι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι συμφωνούν για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τα υλικά αγαθά. Αλλά με την άνοδο του διαδικτύου πολλοί από εμά έχουμε κάπως χάσει το κεφάλι μας. Δεν έχουμε ακόμη καταλάβει ότι πρέπει επίσης να προστατεύουμε όλα τα αγαθά ε, που κυκλοφορούν με ψηφιακά μέσα, μουσική, ταινίες, βιβλία, παιχνίδια βίντεο, λογισμικά το διαδίκτυο δεν θα πρέπει να τετανοποιεί τα πνεύματα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την οποία πρέπει να χαρούμε. Εγγυόμεθα την πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ένα δικαίωμα. Άρα θα πρέπει επίσης σε σχέση με το διαδίκτυο να εφαρμόζουμε τα νομικά κείμενα που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία. Διότι αυτό είναι το δίκαιο. Ή αλλιώ θα έχουμε ζούγκλα, βαρβαρότητα και στη ζούγκλα υπερισχύει ο νόμος του ισχυροτέρου. Ε, αυτό είναι το οποίο επιθυμούμε. Θέλουμε να καταστρέψουμε τον ε, τομέα των ε, δημιουργικών και καινοτόμων επιχειρήσεων με αυτές τις δωρεάν παραχές. Εμείς οι Ευρωπαίοι νομοθέτες θα παραιτηθούμε θα παρασυρθούμε από τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία ή είμαστε ικανοί να σκεφτούμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Σας θέτω το ερώτημα, διότι το αντικείμενο αυτής της έκθεσης είναι ένα σήμα που εκπέμπουμε προς την Επιτροπή για να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις. Ας αφήσουμε τα λαϊκιστικά ανακλειστικά, ας υπερβούμε ε, τις πολιτικάντικες διαμάχες για να εργαστούμε προς το όφελος. να μην αφήσουμε ελεύθερο το πεδίο για την ε, Κομισιόν. Η τύχη των επιχειρήσεων, των δημιουργικών και καινοτόμων και των ατόμων που εξαρτώνται από αυτές είναι στα χέρια μας. Ας μην ξεφύγουμε από το καθήκον μας, η συζήτηση μόλις τώρα αρχίζει. Ευχαριστώ. Τώρα με τη διαδικασία Catch the Eye μπορώ να δεχτώ πέντε ομιλητές. Ορισμένοι που μίλησαν, μίλησαν και στην προηγούμενη ε, συζήτηση, οπότε τώρα θα δώσω το λόγο προς τον κύριο Πιώτα, μάλλον στον κύριο Μπόρις, την κυρία Λίχτεμπέργκερ και στον κύριο Έρενχάουζερ. Τον λόγο έχει ο κύριος Μπόρις καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για αυτή την ε, καλή και ισοσχελισμένη έκθεση η οποία επιβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα τα οποία εξετάζουμε και ε, προβαίνει σε αυτή την προστασία στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο συνάδει με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με, ψηφιακή, με το ψηφιακό πρόγραμμα που πολλές ε, φορές αναφέρεται και σε παρεμφερείς τομείς. Θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή όπως ε, ήδη ανέφερα είναι ισοσκελισμένη και έχει προσόντα διότι δεν αναφέρεται μόνο στην πειρατεία και στην παραποίηση ε, περιοριστικά αλλά προσπαθεί να ε, υποκινήσει μια συνειδητοποίηση των πολιτών οι οποίοι ενδέχεται να μην γνωρίζουν ότι ε, παραβιάζονται τα δικαιώματα άλλων πολιτών και σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση χρειαζόμαστε ένα καλό πρότυπο εμπορίου το οποίο θα προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία, θα προστατεύει τους καινοτόμους και θα επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν εμπορεύματα σε λογικές τιμές Οπότε ε, επανέρχομαι στο σημείο εκκινήξεως αλλά νομίζω ότι το θέμα της πνευματικής ιδιοκλασίας αναφέρεται πολύ καλά και μπορώ, μπορώ να αποδεχτώ την έκθεση. Θα δεχτώ επίσης τον κύριο Ρούμπικ, τον κύριο Γιάρ, την κυρία Ένστρομ και την κυρία Ρόιτοβα η οποία ήταν ε, η συγγήτρια. Έχω μεγαλύτερη δηλαδή και παρακαλώ τώρα τον κύριο Έντσιου να λάβει το λόγο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 πρόκειται για μια γενική ε, πρωτοβουλία του, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στηρίζει αυτή την προσπάθεια και συμφωνώ με την κυρία Γκάλο την εισηγήτρια και θα ήθελα να το είναι σε ορισμένες αρχές οι οποίες θα έπρεπε εμείς να έχουν περιληφθεί. Δηλαδή καταρχήν να υπάρξει μια σαφής διαφοροποίηση και να τονίσουμε την κοινωνικο επι ε, ε, την κοινωνική και οικονομική επίπτωση που θα μπορούσε να έχει η έκθεση αυτή και που μπορεί να έχει ε, σοβαρές επιπτώσεις και η πάροχη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να ενάγονται λόγω των πράξεων των πολιτών τους. Ευχαριστώ κύριος Μάντερς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη συνεργασία της. Η κυρία Γκάλο και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά μαζί μου. Ε, πρόκειται για μία πολύ ε, ζωντανή συζήτηση και πολύ συναισθηματική και στο τέλος παρουσιάστηκε και ένα αναλλακτικό ψήφισμα διότι δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να εγκριθεί το ψήφισμα αυτό. Είναι κρίμα που η συζήτηση ήταν τόσο μεγάλη και παρόλα αυτά δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε λύση. Χρειαζόμαστε περισσότερε καινοτομίε, περισσότερο ηλεκτρονικό εμπόριο, χρειαζόμαστε μια εσωτερική αγορά, αλλά πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, διότι αυτά αποτελούν τη βάση τη καινοτομία. Είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε λύση και ελπίζω αύριο να εγκριθεί το ψήφισμα των φιλελευθέρων. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή έθωση και ελπίζω ο Επίτροπο Μπαρνιέ να μα κάνει μια πρόταση και να παρουσιάσει ένα νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω για τα δικαιώματα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, διότι χρειαζόμαστε άδειε οι οποίες να μην είναι μόνο εδαφικές διότι αυτό αποτελεί απλώς και μόνο ένα πρόστομα επιπλέον. Κυρία Λίχτεμπέργερ, ευχαριστώ. Δεν είναι εύκολο να συμφωνήσουμε εδώ γιατί προσπαθούμε να συνδυάσουμε δύο ασυμβίβατα θέματα. Έπρεπε ίσως να, να, να ασχοληθούμε με την εσωτερική αγορά χωρίς να παρισφρεί το διαδίκτυο που χρειαζόμαστε νέες ε, στρατηγικές που δεν υπάρχουν στο ε, ε, ε, στην νομοθεσία. Επίσης ε, δεν μπορεί κανείς να ξεχνά ότι με το διαδίκτυο επεμβαίνουν νέα στοιχεία στις πληρωμές των πελατών και όταν, όταν απειλούμε με ποινικέ ευθύνες λες και έχω το ένα πόδι ήδη στη φυλακή δεν είναι δυνατόν να προωθήσω και να υποφεληθώ της δυνατότητας της ε, ε, δημιουργικότητας. Οπότε θα πρότεινα να συζητήσουμε πιο ενδελεχώς το θέμα. Αυτό θα ήταν πιο έξυπνο. Ο κύριος Έρενχάουζερ για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καταπολέμηση των παραποιήσεων βεβαίως έχει προτεραιότητα. Πρέπει όμως να σας πω ότι δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω με την έκθεση της συναδέλφου γιατί συμφωνώ με τις ε, επιφυλάξεις διαφόρων νέων ότι στο, 22, στο άρθρο 22 προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εμπόρια στη, ε, στο διαδίκτυο και ε, Επίσης, εις ε, το σημείο αυτό προσπαθούμε να ε, παρεμβάλλουμε μία νομική ασάφισα, ασάφεια. Δεν πρέπει λοιπόν να ποινικοποιήσουμε και να κατηγορούμε εκατομμύρια πολιτών όπως ανέφερε μία προλαλήσεσα και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή οι δομές οι οποίες υπάρχουν ε, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν ε, στο πρόβλημα και θα θέλουν περαιτέρω εξέταση. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ε, ναι κύριε Πρόεδρε, ε, ε περιουσία είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής οικονομίας και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς το θέμα αυτό πρόκειται με ε, ομοφωνία και συνένεση να επιληθεί. Θα είναι πιο απλό για τον ε, καταναλωτή, για τον, ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους μικρούς ιδιοκτήτες να αποκτήσουν άδειες και να ρυθμίσουμε καλύτερα μέσα μέσω αδειών το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρειαζόμαστε ε, μία ε, κοινή ε, αντιμετώπιση της πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι ένα κοινό αγαθό και θα πρέπει οι άδειε οι οποίες χορηγούνται να ισχύσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους πολίτες. Χρειάζεται η αλληλεπίληση αλληλεπίδραση, αλληλεπίδραση και η πολιτική ουδετερότητα για να προχωρήσουμε και βεβαίως χρειαζόμαστε και κυρώσεις για όσους παραβιάζουν το δίκαιο ανταγωνισμού και ε, την νομοθεσία. Ευχαριστώ κυρία, ο κύριος Σίγκστρομ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα με αυτή την έκθεση, αλλά θα επισημάνω ένα βασικό πρόβλημα. Η ασυνέπεια Λέμε στην αρχή ότι δεν έχουμε τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για να νομοθετήσουμε, επομένω θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λάβουμε τα στοιχεία. Και μετά η έκθεση στη συνέχεια προτείνει και επικρίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, διότι δεν έχει προτείνει νομοθεσία και προτείνει νομοθετικά μέτρα στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Συμφωνώ με αυτό που ακούσαμε στην αρχή. Δεν έχουμε τα στοιχεία που, είναι στη... που πρέπει να έχουμε ως ε, αυτοί που χαράσουν την πολιτική. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν έχουν επιτύχει μέχρι τούδε να βρουν μία, ε, μία λύση κατάλληλη για το θέμα. Εγώ ε, υποστηρίζω το ψήφισμα το, ε, της Ενωτικής Αριστεράς, το οποίο λέει να βρούμε πρώτα τα στοιχεία, μετά να σκεφτούμε τι να κάνουμε και μετά να νομοθετήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρ τώρα για ένα λεπτό.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 Ευχαριστώ κύριε Πρέδρε. Οι διαφορετικές ρυθμίσεις στα διάφορα κράτη για την πνευμονική ε, ιδιοκτησία εμποδίζουν την ε, ενιαία προστασία και εμποδίζουν την ε, ενιαία αγορά. Οι παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας πολλές φορές έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και το διαδίκτυο διευκολύνει την κατάσταση. Οπότε η σωστή αυτή η χρησιμοποίηση μπορεί μόνο να προχωρήσει εφόσον υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με σωστές προδιαγραφές για να μπορέσει να ε, ισχύσουν οι αρχές της ευρωπαϊκής αγοράς. Ευχαριστώ και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα ξανασυζητήσουμε πολλές φορές σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και τέλος η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια στην Επιτροπή ΙΠΚΟ για το θέμα αυτό, πρέπει να πω ότι είμαι απογοητευμένη που η συνάδελφος η κυρία Γκάλο δεν έλαβε υπόψη τις συστάσεις μας. Εν τω μεταξύ, ε, σε απάντηση σε δικό μου αίτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το αίτημά μου να δημιουργήσουμε ε, σήματα ευρωπαϊκής πιστοποίησης θα ληφθεί υπόψη ε, Αμέσω. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε το θέμα των παραποιημένων προϊόντων, κυρίω από την Κίνα, μέσω όλων των τρόπων που αναφέρονται στο, στην έκθεση. Είναι κρίμα όμως που προέκυψε τέτοια μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ ε, ευρωβουλευτών ε, για το θέμα ε, των έργων τα οποία είναι αντικείμενο πνευματική ιδιοκτησία και κατεβάζονται από το διαδίκτυο. Δυστυχώ δεν είναι ισορροπημένα τα πράγματα, δεν υπάρχουν σύγχρονοι κανόνε για να δούμε τι γίνεται με του δημιουργού και την προστασία των έργων του. Ε, μάλλον προάγονται τα δικαιώματα αυτών που έχουν τα πνευματικά δικαιώματα ει βάρο και των δημιουργών και των χρηστών. Δυστυχώς η έκθεση ε, δεν μα δίνει την ισορροπία που επιζητούμε. Ευχαριστώ πολύ ε, και τώρα νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ικανοποιήσει του πάντε. Ο κύριο Μπαρνιέ. Ah, Κύριε Πρόεδρε, ακούω πάντα με πάρα πολύ ε, προσοχή αυτά που λένε οι Ευρωπουλευτές. Η Κομισιόν χρειάζεται πάντοτε αυτές τις διαγνώσεις, αυτές τις προτάσεις. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την Μαριέλ Γκαλό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον που εξακολουθεί να επιδεικνύει για το θέμα αυτό και η εισήγηση το αποδεικνύει για τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ξέρω βεβαίω ότι η εισήγηση αυτή υπήρξε αντικείμενο πολλών συζητήσεων, αυτό είναι φυσικό. Νομίζω όμω ότι παρουσιάζει μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα συμφέροντο. Αναφέρομαι στον κύριο Μπόρι και στον κύριο Κιούμπι. όντω μια αποτελεσματική προστασία της πνευματική ιδιοκτησία επιτρέπει να ενθαρρύνουμε την δημιουργικότητα και την καινοτομία, να προστατεύσουμε και τι θέσει εργασία. Αλλά Μιλάμε εδώ για προστασία ε, και δίκαιη ανταμοιβή. Δεν πρόκειται μόνο για την πολιτιστική δημιουργία ή την βιομηχανική δημιουργία. Πέραν αυτών πρόκειται επίσης για μια κάποια ιδέα της ε, δημοκρατίας όταν σκεφτούμε τη δουλειά του δημοσιογράφου που την, στον τύπο ε, πρέπει ε, να αμείβεται και να προστατεύεται καταλήλως. Νομίζω ότι ο κύριος Μπόρις αναφέρθηκε στα προβλήματα υγείας. Ξέρουμε τι κρύβεται γενικά πίσω από τους κινδύνους που σχετίζονται με την παραποίηση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την δέσμευση της Κομισιόν να εργαστεί τους επόμενους μήνες σε στενή συνεργασία με όλες τις ομάδες αυτού του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της πειρατείας και της παραποίησης που ανέφερε κυρία Ρόιτεβες. Θα συνεχίσουμε στην Κομισιό ε, τις αγώνες ε, για να χρησιμοποιώντας νομοθετικά μέτρα, μη νομοθετικά μέτρα και πιστεύω επίσης ότι κάθε αγώνας θα πρέπει να συνοδεύεται με μέτρα θετικά όπως η προώθηση και η ανάπτυξη ε, των προσφορών που είναι θεμητές επιμένω πάνω στην ανάγκη να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών, των νέων, όχι μόνο των νέων, για αυτά τα φαινόμενα χρησιμοποιώντας και αναφέρομαι στον κύριο Άνστρομ χρησιμοποιώντας ανδιαμφισβήτητα στατιστικά στοιχεία για τις συνέπειες και το εύρος και τη σημασία της παραποίησης και της πειρατείας και με την όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση για τις συνέπειες πάνω στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό ανέφερε ο κύριος Σαντσού προηγουμένως. Η Κομισιό θα αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη του παρατηρητηρίου και των άλλων μέτρων που αναγγέλθηκαν στην ανακοίμνωσή μας του Σεπτεμβρίου 2009 προς την διοικητική συνεργασία και διάλογο δια βιομηχανικό. Θα παρουσιάσω ε, το φθινόπορο αυτά τα θέματα παραποίησης, όλες τις διαστάσεις της παραποίησης και ε, της πειρατείας που θα συνοδεύεται με ένα σχέδιο δράσης που θα βασίζεται συγκεκριμένα προς την έρευνα και την επικοινωνία, ως προς την κατάρτιση, την εκπαίδευση προσωπικού στις χώρες μας, ε, στον έλεγχο των συνόρων θα βασίζεται στις εργασίες και στην πραγματογνωμοσύνη του παρατηρητηρίου που θα θεσπίσουμε με τρόπο αξιόπιστο και συγκεκριμένο. Επίσης αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση ε, του νομοθετικού πλαισίου για την σεβασμό και προστασία της πνευματική ιδιοκτησίας θα πρόκειται βεβαίως για ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό. Η λύση θα βασίζεται σε μια ισορροπημένη αναλογική ε, πρόσβαση προστατεύοντας τα δικαιώματα ε, των ε, καταναλωτών και θα ήθελα να πω στην κυρία Λισβερζέ ότι δεν πρόκειται να ποινικοποιήσουμε ορισμένε συμπεριφορέ κυρίω των νέων. Όχι, όχι, δεν πρόκειται γι' αυτό. Η Κομισιό ετοιμάζει για το φθινόπωρο μια έκθεση για την Οδηγία 2004-48 EC σχετικά με τον σεβασμό της, ιδιοκ... της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και το λέω στον κύριο Έντελς και στην κυρία Γκαλό που επέμεινε πάνω σε αυτό το σημείο βάσει της έκθεσης αυτής θα προτείνουμε όπως νομίζω ότι αυτό θα καταστεί αναγκαίο τροπολογίες σε αυτό το κείμενο για να βελτιώσουμε την προστασία των ε, δικαιωμάτων αυτών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε την κυρία Γκάρλο και τους συναδέλφους. Αύριο ψηφίζουμε στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερίδια διάταξη είναι η έκθεση του Ζωάου Φερέιρο για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Και να δώσω το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Κύριε Φερέιρα, έχετε το λόγο.